Bueno, eh, decía Έλεγα προηγουμένως θα ήθελα να καλωσορίσω τους δύο εμπειρογνώμονες που κάλεσε η κυρία Γιώτοβα στη σημερινή μας συνεδρίαση που θα μας δώσουν πιο συγκεκριμένες πληροφορίες το θέμα που μας απασχολεί που είναι οι αληφτικές δραστηριότητες και η μελλοντική διεχείριση στο στον Εύξηνο Πόντο. Καλωσορίζω λοιπόν τον κύριο Βιολίν Ράικοφ του Οικενογραφικού Ινστιτούτου της Βουλγαρίας και τον κύριο Γιορτάν Κοσποντίνοφ, διευθυντή τη... υπεύθυνο της ε, Ένωσης ε, Αλληλευτικών Προϊόντων Θα δώσουμε το λόγο στην κυρία Γιώτοβα πρώτα μετά για 10 λεπτά στον καθένα τους δύο εμπειρογνώμονες και μετά θα ανοίξω η ζήτηση. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θα είμαι πάρα πολύ σύντομη. Πρόκειται για την δεύτερη ανταλλαγή απόψεων που αφορά την πρόταση πρωτοβουλία, την έκθεση πρωτοβουλίας για την τρέχουσα και μελλοντική διαχείριση αλίας στον Ευξηνοπόντο. Δεν θα μπω σε λεπτομέρειες. Ήδη της είχα κάνει μια πρώτη παρουσίαση τον προηγούμενο μήνα. Θα ήθελα να πω δύο λόγια για τους προσκεκλημένους μας από την ε, Βουλγαρία. Ο κύριος Ράικοφ είναι ένας από τους καλύτερους βιολόγους. Γνωρίζει πάρα πολύ καλά τα αλλιευτικά αποθέματα. Εργάζεται... Ε, στο Ινστιτούτο στο Κενογραφικό Ινστιτούτο μας. Ο κύριος Γιορτάν Γκοσποντίνοφ εκπροσωπεί την Ένωση Παραγωγών ε, Προϊόντων Αλίας Big Fish και εκπροσωπεί τους αλίες της Βουλγαρίας στη Μαύρη Θάλασσα. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω που επιτρέπετε να παρουσιάσετε την έκθεση αυτή στα πλαίσια κοινή αλλιευτικής πολιτικής ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση θα ήθελα αν θέλετε να δώσουμε το λόγο στον κύριο Ράικο. ευχαριστώ λέει πρόεδρος. Ξέρω ότι πολλού ε, συναδέλφου του ενδιαφέρουν πολλά άλλα θέματα. Δεν θέλουμε να χάσουμε χρόνο. Θα δώσω πρώτα απ' όλα το λόγο στον κύριο Ράικοφ. Έχετε το λόγο. Περίπου 10 λεπτά σας δίνω, λέει η Πρόεδρο. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι, κυρίες και κύριοι εκπρόσωποι Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της Επιτροπής ε, στον τομέα της αλίας και σε θέματα σχετικά με την βιοπικιλότητα θα ήθελα να σας πω ότι υπάρχουν στην περιοχή της Μαύρης Θάλασσα τρεις συμβάσεις. Πρέπει να σας πω ότι από θεσμικής πλευράς η κατάσταση έχει ως εξής. Όλες οι χώρες είναι συμβαλόμενα μέρη της Σύμβασης του Βουκουρεστίου, τέσσερι είναι συμβαλόμενα μέρη της ε, Συμφωνίας για την προστασία των ε, των κοιτοειδών στην Μαύρη Θάλασσα, την ε, ε, Μεσόγειο και στην περιοχή του Ατλαντικού και οι προσπάθειες τις οποίες κάνουμε στα πλαίσια της Επιτροπή μας είναι να προσπαθήσουμε να διασφαλίσουμε τους ζώντες αλλιευτικούς πόρους και να... Και έχουμε σημαντικά επιτεύγματα ε, από το 2008-2009 και μετά. Υπάρχουν, πρέπει να σας πω, μεγάλες διαφορές ε, μεταξύ των διαφόρων χωρών και έλλειψη συντονισμού σαν αφορά την αλληλεία. Ε, γίνονται προσπάθειες ώστε να μην επιδεινώνονται τα αποθέματα των αλλιευτικών ειδών και να μην υπάρχει υπεραλληλία στην περιοχή. οι προσπάθειες που θα πρέπει να γίνουν πρέπει να γίνουν για να αποφευθεί η υπεραλίευση και να μην ε, μειωθούν τα αλλιεύματα τα οποία υπάρχουν στην Μαύρη Θάλασσα. Γι' αυτό θα πρέπει να εφαρμοστεί μια πολιτική διαχείριση της αλλίας. Γενικά η διαχείριση των αλλιευτικών πόρων ε, είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να γίνει με την στοχοθέτηση. Η αλία είναι ένας πάρα πολύ σημαντικός οικονομικός παράγοντα για τη μαύρη θάλασσα. Η κατανάλωση ε, των αλλιευτικών ειδών τα τελευταία χρόνια έχει αυξηθεί κατά 50%. Υπάρχει και ε, πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για συνεργασία σε επίπεδο διασυνοριακό. Θα πρέπει να υπάρχουν κοινά ωφέλη για όλες τις χώρες και σωστή ενημέρωση για τις δραστηριότητες στην περιοχή. Η διαχείριση λοιπόν της αλίας είναι ένα θέμα προτεραιότητας για μας. Πρώτα απ' όλα θα πρέπει να δούμε το θέμα της υπεραλίας θα πρέπει να δούμε πώς θα εισαγάγουμε νέα είδη, πώς θα προστατεύσουμε τους ε, οικισμούς. Προσπαθώ να είμαι σύντομο. Τα προβλήματα τα οποία θέλουμε να ξεπεράσουμε είναι να ε, δούμε πώς θα καθορίσουμε την παραγωγικότητα και τα είδη των αλλιευτικών πόρων να δούμε ποιες είναι οι μέθοδοι εκμετάλλευσης ώστε να διαχειριστούμε σωστά την παραγωγικότητα, να εξετάσουμε και να αξιολογήσουμε τις ε, διάφορες εναλλακτικές λύσεις για την διαχείριση και την κατανομή των όφελων, να μην καταστρέφουμε τους οικισμούς, να δούμε πώς θα βοηθήσουμε τις, ε, τα επαπειλούμενα είδη, πώς θα βελτιώσουμε την διαχείριση των προστατευόμενων περιοχών, πώς θα μπορέσουμε να διαχειριστούμε αφού καθορίσουμε πρώτα τις διασυνεργασιακά προστατευόμενες περιοχές και να αποκαταστήσουμε την ε, κατάσταση σε κάποιες περιοχές οι οποίες έχουν υποστεί βλάβες. Γι' αυτό θα πρέπει να υπάρχει πολιτική βούληση, θέσπιση των κατάλληλων μηχανισμών και συστημάτων διαχείρισης. Πιστεύω ότι θα πρέπει να γίνει πρώτα απ' όλα η αξιολόγηση όλων των μεθόδων για την προστασία όλων των αλλιευτικών πόρων, γιατί αυτό είναι κάτι το οποίο δεν έχει γίνει σωστά μέχρι τώρα. Οι επιπτώσεις των κλιματικών αλλαγών επίσης είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να μελετήσουμε και η μελέτη της θερμοκρασίας των οικοσυστημάτων επίσης και η σημασία τους για την αλληλεία να μελετηθούν. Επίσης θα πρέπει να δούμε πώς θα προστατεύσουμε τους ζώντες ε, θαλάσσιους πόρους και θα κάνουμε σωστή αλληλεία χωρίς να μειώσουμε τη, τους αλληλευτικούς πόρους. Με σωστή διαχείριση λοιπόν θα πρέπει να βελτιώσουμε το σύστημα που υπάρχει. Ευχαριστώ σας. Ευχαριστώ. Και τώρα το λόγο έχει ο κύριος Γκοσποντίνοφ. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, μέλη της Επιτροπής Αλίας, του Συμβουλίου της Επιτροπής. Θα προσπαθήσω να είμαι σύντομος ο συνδυασμό ο, η ένωση των παραγωγών ε, και παραγωγών της περιοχής της Μαύρης Θάλασσας Big Fish, BG Fish δεν να σας παρουσιάσει κάποιους από τους ε, στόχους. Εδώ η Μαύρη Θάλασσα καταρχήν έχει επικοινωνία με άλλες ε, θαλάσσιες περιοχές όπως παραδείγματο χάρη το Βόσφαιρο. Υπάρχουν επίσης οι ποταμοί που φτάνουν μέχρι τη Μαύρη Θάλασσα με όλες τις συνέπειες. Η Μαύρη Θάλασσα επηρεάζεται λοιπόν από όλες αυτές τις ε, θαλάσσιες οδούς με πολλούς τρόπους. Υπάρχουν και άλλες λεκάνες στις οποίες υπάρχουν παρόμοια προβλήματα. Θεωρώ ότι ιδιαίτερη σημασία πρέπει να δοθεί σε αυτές τις ε, λεκάνες, όχι μόνο στην Μαύρη Θάλασσα, αλλά και στις γειτονικές περιοχές. Όταν μιλώ για ειδική προσοχή, ενώ υπεύθυνη πολιτική που να βασίζεται στα χαρακτηριστικά αυτής της περιοχής, της Μαύρης Θάλασσας και την προστασία των ειδών που ζουν στη Μαύρη Θάλασσα. Μια ειδική πολιτική, η οποία θα πρέπει να συνδυάζεται και με πολιτιστικά μέτρα, και όχι μόνο οικονομικά, που θα πρέπει να είναι μία από τις ε, προτεραιότητες όσον αφορά την παρούσα και μελλοντική διαχείριση των αληθικών πόρων της Μαύρης Θάλασσας. Η υλοποίηση αυτής της πολιτικής στη Μαύρη Θάλασσα, της IMP, αλλά και η επέκταση των ε, βέλτιστων πρακτικών, η εμπειρία που έχουμε από τη Βαλτική θάλασσα θα πρέπει να εφαρμοστούν εκεί που μπορούν στην ε, Μαύρη θάλασσα. Στη χώρα μας έχουμε μια πολιτική όσον αφορά τον τουρισμό και την αλία που βεβαίως πάντα δεν εφαρμόζεται σε άλλα γειτονικά κράτη. 2.000 άτομα εργάζονται και επηρεάζονται από την αλία στην περιοχή αυτή στις παράκτιες περιοχές, 2.000 σκάφη και... και 25 επιχειρήσεις οι οποίες δραστηριοποιούνται σε μικρές ε, πόλεις ε, και χωριά όπου Οι οικονομικές συνέπειες αυτή τη δραστηριότητα είναι καθοριστικέ για τους κατοίκους της περιοχής αυτής. Οι αλληλεί αυτοί συνήθως ε, δεν έχουν άλλες εναλλακτικές ε, πηγές οικονομικές δραστηριότητες και η ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική θα πρέπει να βρει λύσεις για τα προβλήματα αυτών των περιοχών. Πρώτον, τα θαλάσσια σαλιγκάρια και ο πολλαπλασιασμός τους που απειλεί άλλες, άλλα είδη όπως παραδείγματος χάρη τα λευκά και μαύρα μύδια. Όπως ξέρετε, τα στρίδια της Μαύρης Θάλασσας είναι είδος υποεξαφάνιση. Και αυτό διότι απειλούνται από τα θαλάσσια σαλιγκάρια. Έχουν πολλαπλασιαστεί λοιπόν αυτοί οι οργανισμοί και θα πρέπει να βρούμε εναλλακτικές μεθόδους αλλιώς που να μην καταστρέφουν το υπέδαφος και το βυθό της θάλασσας. Όχι μόνο δηλαδή με το υποβρύχιο ψάρεμα και να βρεθούν εναλλακτικές μέθοδοι. Επί αρκετά χρόνια υπήρξαν ε, αμφισβητήσεις όσον αφορά την υλοποίηση εδώ της κοινοτική νομοθεσίας και μόνο έξι γειτονικά κράτη ανήκουν στην ε, Ευρωπαϊκή Ένωση, κάτι που σημαίνει ότι πολλές φορές δεν έχουμε ακριβή και αξιόπιστα στοιχεία όσον αφορά την αλληλευτική δραστηριότητα στην περιοχή. Χρειάζεται μια κοινή πολιτική μεταξύ των έξι γειτονικών χωρών και για λόγους οικολογικούς για την προστασία της Μαύρης Θάλασσας, αλλά και για οικονομικούς λόγους. Η κοινή συμφωνία μπορεί εδώ να αντικατασταθεί από ένα, ε, μια συμφωνία πλαίσιο. Επίσης δεν υπάρχει συστηματική και επιστημονική πληροφόρηση όσον αφορά την Μαύρη Θάλασσα. Βεβαίως Υπάρχουν πολλές δυνατότητες ε, στα δύο επιστημονικά Ινστιτούτα. Πιστεύουμε ότι επιστήμονες, εμπειρογνώμονες από την Ευρώπη και από κράτη που δεν ανήκουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να συνεργαστούν. Δεν υπάρχει αρκετή ενημέρωση, δεν υπάρχουν αρκετά στοιχεία και πληροφορίες για τη Μαύρη Θάλασσα, τα είδη που βρίσκονται σε αυτήν και την ίδια ώρα έχουν επιβληθεί ποσοστώσεις για τα υποεξαφάνιση ήδη πιστεύουμε ότι δεν έχουμε αξιόπιστα στοιχεία και θα πρέπει οπωσδήποτε να χρησιμοποιήσουμε και την τεχνογνωσία της, του συνδέσμου μας και των μελών της ε, BGFISH. Οι αλείς γνωρίζουν την περιοχή αυτή, γνωρίζουν τη Μαύρη Θάλασσα, γνωρίζουν πού βρίσκονται τα διάφορα είδη, γνωρίζουν τις ιδιαιτερότητες, τις εποχές. Χρειάζεται λοιπόν να δημιουργηθεί ένας οργανισμός διαχειριστικός για την Μαύρη Θάλασσα με ρόλο συντονιστικό και να καθοδηγηθεί μια επιτροπή επιστημόνων με σκοπό να ελοποιηθεί τελικά μια πολιτική για την προστασία των απειλούμενων ειδών και αυτό βεβαίως θα πρέπει να ακολουθείται και από ένα πολιετές πρόγραμμα όσον αφορά τη διαχείριση των αποθεμάτων στο οποίο θα συμμετάσχουν όλα τα κράτη της Μαύρης Θάλασσας. Η Βουλγαρία προσχώρησε στην Ευρωπαϊκή Ένωση αργά και δεν μπορέσαμε να υποφεληθούμε από την στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την αντικατάσταση του στόλου μας. Τουλάχιστον ε, σε σχέση με άλλους στην Μαύρη Θάλασσα. Αντιμετωπίζουμε σήμερα λοιπόν την πραγματικότητα με περιορισμούς που όπως καταλαβαίνετε δύσκολα γίνονται αποδεκτοί από τους αλλοίς και η κοινή αλληλευτική πολιτική δύσκολα αν θέλετε γίνεται αποδεκτή από τους αλλιείς. Είναι δύσκολο να διαπραγματευτεί κανείς ε, με τη φύση. Γι' αυτό και χρησιμοποιούμε και τους μη κυβερνητικούς οργανισμούς ε, στην περιοχή. Χρειαζόμαστε περισσότερη ανάπτυξη και ευημερία προς όφελος όλων όσων ζουν και εργάζονται στην περιοχή της Μαύρης Θάλασσας. Προστασία των ειδών και ιδιαίτερα όσον αφορά προϊόντα τα οποία είναι προϊόντα με υψηλή διατροφική αξία. Σας ευχαριστώ πολύ. Θέλει κανείς το λόγο παρακαλώ, κυρία Λόβιν. Uh, Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω και τους δύο για την ενδιαφέρουσα παρουσίαση. Είμαι Σουηδέζα. Είναι παράκτια χώρα της Βαλτικής. Όλα όσα είπατε ε, χτυπούν κάποιο καμπανάκι μέσα μου. Ε, η Βαλτική είναι μια υφάλμηρη θάλασσα, είναι κλειστή λεκάνη και έχουμε αντίστοιχα προβλήματα ε, εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Αλλά τώρα αρχίζουμε να κινούμαστε προς τη σωστή κατεύθυνση στη Βαλτική. Και νομίζω ότι αυτό έγινε χάρη πολλών εξεχεριών. Προσπαθήσαμε να επιτύχουμε μια διεθνή συμφωνία μεταξύ των κρατών που είναι παράκτιες στη Βαλτική. Ε, σας άκουσα πραγματικά με έκπληξη ακούγονται ότι δεν έχετε κανένα διαχειριστικό φορέα στη Βαλτική θάλασσα. Δεν έχουν κανένα πιο φορέα τα παράκτια κράτη της Μαύρης θάλασσας. Νομίζω ότι είναι πραγματικά ανησυχητικό. Είναι ανησυχητικό το, το ότι δεν υπάρχει καν συνεργασία. Ε, δεν ανταλλάσσεται επιστημονικά στοιχεία για τη Μαύρη θάλασσα. Ε, θα ήθελα να σας συγχαρώ που έχετε ακόμα ψάρια στη Μαύρη θάλασσα. Γιατί χωρίς τέτοιες ε, κινήσεις ε, θα οδηγηθείτε σε καταστροφή. Ήθελα να σα το πω αυτό. Δεν έχω συγκεκριμένε ερωτήσεις. Έχετε να κάνετε πάρα πολλή δουλειά και ελπίζω η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, να σας υποστηρίξει. Εμείς βεβαίω θα σας υποστηρίξουμε όσο μπορούμε για την δημιουργία αυτών των φορέων που είναι εκ των όνου κάνευ αν θέλουμε να υπάρξει διαχείριση οποιασδήποτε θαλάσσια λεκάνης. Ευχαριστώ. Μάλιστα. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα καταρχάς να συγχαρώ την κυρία Γιάτοβα για την πρωτοβουλία της πρόκειται, για σημαντική πρωτοβουλία. Θα ήθελα να συγχαρώ τους δύο εισηγητές για τις εξηγήσει που μας έδωσαν. Και να πω το εξή: Το πρώτο πρόβλημα το οποίο υπάρχει κατά την άποψή μου και πείτε μου την άποψή σας είναι το θέμα της διαχείρισης δεν μιλώ για τις ε, σχέσεις που μπορείτε να έχετε με τις γειτονικές σας χώρες, αλλά υπάρχει κάποια πολιτική διαχείριση, διακυβέρνηση των ληφτικών πόρων. Μιλήσατε βεβαίως για το ότι σας ενδιαφέρει να μειώσετε το μέγεθος του αλληλευτικού στόλου. Ξέρουμε ότι υπάρχουν πάρα πολλά σκάφη τα οποία αλληλεύουν. Ποιος είναι ο στόχος που θέλετε να υλοποιήσετε. Η κυρία Ράντοστ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να σε ευχαριστήσω και τους δύο για όλες τις πληροφορίες, τρομερά ενδιαφέρουσες. Θα ήθελα κυρίως να ευχαριστήσω την ε, συναδελφό μου, την κυρία Ιώτοβα, γιατί αν δεν είχε λάβει αυτή την πρωτοβουλία, νομίζω ότι δεν θα είχαμε καμία ιδέα για το τι συμβαίνει στη Μαύρη Θάλασσα. Γι' αυτό πραγματικά την ευχαριστώ θερμά. Συμφωνώ με αυτά που είπατε κυρία Λέβιν. Ε, χρειάζεται πραγματικά πρωτοβουλίες, χρειάζεστε δράση. Γιατί αν δεν ρυθμίσετε τα πράγματα το συντομότερο δυνατόν, θα αντιμετωπίσετε σοβαρότατα προβλήματα ανάλογα με αυτά που αντιμετωπίζουν άλλες περιοχές και κάποια στιγμή θα βρεθείτε χωρί ψάρια. Ε, μιλήσατε για ένα σαλιγκάρι το οποίο ε, είναι χωροκατακτητικό. Θα ήθελα να μου πείτε ποιες είναι πρωτοβουλίες που θέλετε να αναλάβετε, ούτως ώστε να ε, σταματήσετε από τον πολλαπλασιασμό αυτών των σαλιγκαριών. Ε, δεν νομίζω ότι είναι από τη μαύρη θάλασσα το σαλιγκάρι, αλλιώς δεν θα είχαμε αυτό το πρόβλημα. Ε, και εμείς έχουμε αντίστοιχα προβλήματα στη μαύρη θάλασσα στην ε, Βόρεια Θάλασσα, συγγνώμη. Τι σκοπεύετε λοιπόν να κάνετε. Να σας ευχαριστήσω για την πολύ ενδιαφέρουσα παρουσίαση. Πρόκειται για τη δεύτερη έκθεση που αφορά την Μαύρη Θάλασσα και πολύ σωστά είπατε νομίζω και οι δύο ότι η κατάσταση είναι δύσκολη. 16 κράτη γύρω από τη Μαύρη Θάλασσα και μόνο ελάχιστα στην ε, Ευρωπαϊκή Ένωση. Δύο. Συμμετέχουν στην ε, κοινή πολιτική μόνο έξι. Μόνο έξι. Α, έξι όχι οι δύο. Για μια αηφόρο ανάπτυξη τουλάχιστον να εγγυθούμε ότι στο μέλλον θα υπάρξει κάποια τέτοια, θα πρέπει να συμμετέχετε, να συνεργαστείτε με τα άλλα τέσσερα κράτη. Δεν ξέρω, η Τουρκία ας πούμε που έχει μια μεγάλη ακτή στο νότο συνεργάζεται με τη Βουλγαρία. αυτά τα 12 μίλια υπάρχουν συμφωνίες ότι δηλαδή μπορεί κανείς να μπει τρία μίλια και να ψαρέψει δεν ξέρω υπάρχει αυτή η συμφωνία που ισχύει παντού γιατί ξέρω ότι αυτή η εγγύηση δίνεται τα περισσότερα κράτη εδώ και χρόνια. Με την Ουκρανία παραδείγματο χάρη, με τη Ρωσία. Πώς ε, συνεργάζεστε και βέβαια τα υπόλοιπα ανατολικά κράτη. Eh, Θα ήθελα κι εγώ να πω το εξής. Η Μαύρη Θάλασσα δεν είναι μέρος της ε, ε, του Κοινού Συμβουλίου της Αλίας ε, για την Μεσόγειο. Υπάρχει ο Ναι, ναι, σωστά το είπε. Ευχαριστώ. Να επαναλάβω αυτό που είπα τελευταία φορά, ότι καλωσορίζουμε την πρωτοβουλία της κυρίας Γιώτοβα, πρωτοβουλία που υλοποιείται με αυτή την έκθεση και συμμεριζόμαστε την ανησυχία ότι Υπάρχει σοβαρή και αδύρυτη ανάγκη να κάνουμε κάτι στη Μαύρη Θάλασσα. Και καλωσορίσω φυσικά την έκθεση των δύο εμπειρογνωμόνων. Ε, σε μεγάλο βαθμό συμφωνούμε με την αξιολόγηση που έγινε για την κατάσταση των πόρων στη Μαύρη Θάλασσα και για τα μέτρα που είναι απαραίτητα για να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα. Λοιπόν, το βασικό θέμα είναι η περιφερειακή συνεργασία, γιατί όπως είπατε όλοι σας, η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι παρούσα μόνο με δύο κράτη-μέλη στη Μαύρη Θάλασσα και υπάρχει ανάγκη για να δημιουργηθεί διάλογος με άλλες χώρες της Μαύρης Θάλασσας, ούτως ώστε να προχωρήσουμε στο διάλογο για να συζητήσουμε τα θέματα καλύτερων ε, επιστημονικών συμβουλών. Ε, ένας επιστήμονας από τη Ρωσία και την Ουκρανία και την Τουρκία συμμετείχαν ε, στη τεχνική αυτή και επιστημονική επιτροπή. Ε, θα ξαναγίνει το ίδιο φέτος. Αναφέρεται επίσης το πρόβλημα των θαλάσσιων σαλιγκαριών. Με βάση τα όσα είπε η Επιστημονική και Τεχνική Επιτροπή, θα δώσει φέτος συμβουλές, γιατί το ζητάμε εμείς για το θέμα αυτό της αντιμετώπισης του σολυγκαριού. Είναι η πρώτη απόπειρα να αντιμετωπιστεί το θέμα από την Τεχνική και Επιστημονική Επιτροπή. Σωστά είπατε ότι υπάρχουν τρεις ε, συμβάσεις οι οποίες ρυθμίζουν ε, τη διαχείριση των πόρων στη Μαύρη Θάλασσα. Α, συγγνώμη. Η σύμβαση του Βουκουρεστίου ασχολείται με τη ρήπανση της Μαύρης Θάλασσας η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι συμβαλόμενο μέρος αυτής της σύμβασης. Ε, ζητήσαμε να γίνουμε μέρος, μέλος και μας υποστήριξε βέβαια η Βουλγαρία και η Ρουμανία, αλλά η Ρωσική Ομοσπονδία μας το αρνήθηκε, τουλάχιστον μέχρι στιγμής έτσι είναι τα πράγματα. Όπως είπε και μία συνάδελφος, το GFCM έχει αρμοδιότητα για τη Μαύρη Θάλασσα επίσης. Προτείνω το εξή. Δεν αποκλείουμε να γίνουν κάποιε συζητήσει, να ανταλλαγούν κάποιες σκέψεις για να δούμε αν μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα ειδικό οργανισμό για τη Μαύρη Θάλασσα. Αλλά πέραν αυτού θα πρέπει να αρχίσουμε τις εργασίε μας στα πλαίσια του GFCM, όπου έχουμε διάφορες χώρες, διάφορα συμβαλόμενα μέρη παρόντα και έχουμε λάβει και μηνύματα από τη Ρωσική Ομοσπονδία ότι μπορεί να ενταχθεί και αυτή στην GFCM. Θα έχουμε την Τουρκία λοιπόν και τη Ρωσία στο GFCM. Μπορούμε να ξεκινήσουμε το GFCM και να συνεχίσουμε τις συζητήσεις για να δούμε αν σε κάποια φάση μπορούμε να οδηγηθούμε στη δημιουργία ενός ειδικού οργανισμού για την ε, Μαύρη Θάλασσα. Μην ξεχνάτε ότι μία περιφερειακή οργάνωση Αλλία για να δημιουργηθεί χρειάζεται πάρα πολύ χρόνο. Επομένω, εμεί θα πρέπει να δουλέψουμε τώρα με αυτά που έχουμε στα χέρια μα. Επίση, αρχίσαμε το διμερή διάλογο με άλλε χώρε τη Μαύρη Θάλασσα. Η κυρία Δαμανάκη πήγε στην Τουρκία και στην ε, Ρωσία τον Οκτώβριο και τον Δεκέμβριο, αν αναπατώμε στις ημερομηνίες. Ε, σε επίπεδο υπηρεσιών μα, συζητήσαμε πριν από δύο εβδομάδε με Ρώσου ομολόγου μα στα πλαίσια του Μνημονίου κατανόηση για την Αλία. Και η Μαύρη Θάλασσα ήταν στη ημερήσια διάταξη. Αρχίσαμε λοιπόν τη συζήτηση για τη Μαύρη Θάλασσα και με του Ρώσου. Θα έχουμε μια συνάντηση στο τέλο του μήνα με την Τουρκία επίσης, ε, όπου θα μιλήσουμε για το πρόβλημα της ε, διαχείριση Αλία στη Μαύρη Θάλασσα και τη Μαύρη Θάλασσα εν γέννη. Η πρόθεση τη κυρία Δαμανάκη είναι να αρχίσει ένα διάλογο με τι άλλε χώρε και κυρίω με την Ουκρανία πριν από το τέλο του 2011 όπως είπα και με την Ουκρανία, που είναι μία από τις σημαντικές ε, χώρες που αλλιεύουν ε, στη Μαύρη Θάλασσα. Πολύ σύντομα λοιπόν, αυτές είναι οι πληροφορίες που ήθελα να σας ε, κοινοποιήσω. Έχουμε ξεκινήσει τη δουλειά, είμαστε πιο δραστήριοι πια. Επίσης, εξετάζω μια στρατηγική ε, ολοκληρωμένης θαλάσσιας πολιτικής για τη Μαύρη Θάλασσα. Μία από τις προτεραιότητες θα είναι σίγουρα η αλία και η διαχείριση της αλίας. Υπάρχουν θέματα θαλάσσιας ασφάλειας στην περιοχή. Blue. Προς το παρόν, αυτό γίνεται μόνο σε επίπεδο υπηρεσιών. Έχουμε ξεκινήσει να δουλεύουμε σε επίπεδο υπηρεσιών της Κομισιόν δηλαδή, αλλά έχουμε ξεκινήσει και διάλογο με χώρες της ε, Μαύρης Θάλασσας. Θα θέλαμε επίσης να επωφεληθούμε ε, της ευκαιρίας ε, λόγω της Προεδρίας της Ρουμανίας ε, της Επιτροπής Μαύρης Θάλασσας και να επωφεληθούμε από, ίσως να προχωρήσουμε διάφορες πρωτοβουλίες. Ξεκινάμε λοιπόν το διάλογο, ούτω ώστε από τη μία να βελτιώσουμε την επιστημονική γνώση, τις επιστημονικές συμβουλές και από την άλλη να δημιουργηθεί ένα πλαίσιο για να υπάρξουν μέτρα διαχείρισης για τη Μαύρη Θάλασσα. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Θα δώσω τώρα το λόγο στους δύο προσκεκλημένους και θα ολοκληρώσω τη συζήτηση κυρία Ιώτοβα. Σα δίνω το λόγο για να απαντήσετε στις ερωτήσεις που τέθηκαν. Κύριε Ράικοφ, πρώτα απ' όλα εσείς και μετά ο κύριος Γκοσποντίνοφ. Κύριος Ράικοφ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Το ενδιαφέρον της Μαύρης Θάλασσας είναι φυσικά αυτή τη στιγμή για σας είναι η αλία. Εκεί εστιάζεστε. Ε, μιλήσατε για τη συμμετοχή χωρών στο GFCM. Πριν από λίγες εβδομάδες ε, συμμετείχα στις εργασίες της Επιστημονικής και Τεχνικής Επιτροπής του GFCM ως σημείο επαφής. Και με έκπληξη σημείωσα την παρουσία παρατηρητών από τη Ρωσική Ομοσπονδία για πρώτη φορά, που εξέφρασαν τη θέλησή τους να κάνουν κάθε προσπάθεια, ούτως ώστε να δημιουργηθεί κάποιος περιφερειακός οργανισμός, ειδικά για την αλία. για τις συζητήσεις που έλαβαν χώρα σε αυτή την ε, Επιτροπή. Η πιο σημαντική, το πιο σημαντικό θέμα είναι ότι όλες οι χώρες που ήταν παρούσες ως χώρες επαφής ή ως παρατηρήτριες συμφωνούν Θέλουμε λοιπόν να δημιουργήσουμε μια περιφερειακή επιτροπή με ομάδες εργασίας και υποομάδες εργασίας, όπως ακριβώς το GFCM. Και λόγω των συγκεκριμένων θεμάτων που είναι διαφορετικά από την Μεσόγειο, θα πρέπει οι επιστήμονες της Μαύρης Θάλασσας να δημιουργήσουν δική τους περιφερειακή ε, επιτροπή. Αυτά όσο ό,τι αφορά το GFCM. Σε ό,τι αφορά τα τάκ και τις ποσοστώσεις, από το 2007 μόνο η Βουλγαρία και η Ρουμανία έχουν ε, ε ποσοστώσεις για το, τη σαδελόρεγγα, μικρά, δηλαδή μικρό πελαγικό είδος. Επίσης θα, έχουμε και, θα συμπεριλάβουμε και κάποια καρκινοειδή. Ο άλλος ομιλητής. Με μεγάλη χαρά άκουσα ότι εκφράζετε, εκφράζετε και εσείς ανησυχίες, όπως και εμείς, για τα όσα συμβαίνουν στη Μαύρη Θάλασσα, πρέπει να υπάρχει ενεργή συμμετοχή. Σε πολιτικό επίπεδο και συμμετοχή από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Χρειαζόμαστε ένα συγκεκριμένο έγγραφο. Η Μαύρη Θάλασσα είναι η διάζουσα περίπτωση. Και το να εμπλέξουμε τα άλλα παράκτια κράτη ε, σε ένα πειραματισμό υψηλού επίπεδου θα δημιουργήσει προσδοκίες για το μέλλον. Σε ό,τι αφορά αυτό το χωροκατακτητικό είδος που είναι το θαλάσσιο σαλιγκάρι και τα, μέρη, και τα μέτρα που μπορούμε να λάβουμε, έχουμε κάποια, κάποιες ιδέες, αλλά χρειαζόμαστε επιστημονικά στοιχεία και έρευνα για αυτό το θέμα. Θα χρησιμοποιήσουμε λοιπόν αυτό που, αυτή την πρόταση που έκανε η εκπρόσωπος της Επιτροπής για τα σαλιγκάρια Ξέρουμε ότι πρέπει να γίνει μια ανάλυση πολύ λεπτομερής για να βρούμε την καταλληλότερη μέθοδο για να τα πιάνουμε αυτά τα σαλιγκάρια, ούτως ώστε να μην βλάπτουμε το οικοσύστημα της ε, Μαύρης Θάλασσας και για να διαφυλάξουμε το βιωτικό επίπεδο των ανθρώπων της Μαύρης Θάλασσας που ζουν από αυτή τη δραστηριότητα. Σας ευχαριστώ κυρία Ιώτοβα. Δύο λόγια από μένα για να τελειώσουμε. Θα ήθελα να σα ευχαριστήσω, κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ όλου του συναδέλφου που πήραν μέρο στη συζήτηση. Σα ευχαριστώ για τη δέσμευσή σα. Ε, σα ευχαριστώ που καταλαβαίνετε τη σημασία του θέματο. Ξέρετε ότι υπάρχουν ποικίλα θέματα που απασχολούν τη Μαύρη Θάλασσα. Το βασικό πρόβλημα είναι ότι δεν υπάρχει έρευνα βάσιμη. Ε, γιατί δεν υπάρχει συμφωνία μεταξύ των έξι παρακτήων χωρών. Η έκθεση η οποία θα εκδοθεί θα σας δώσει κάποιες ιδέες για το πώς να υπάρξει έρευνα για τα θέματα που απασχολούν τη Μαύρη Θάλασσα πριν δημιουργηθεί ένας νέος φορέας. Όσο περισσότερο το συζητάμε, τόσο περισσότερο είμαι πεπισμένο ότι χρειαζόμαστε κάποια οργάνωση, κάποιο φορέα. Γιατί η Μαύρη Θάλασσα πραγματικά είναι ιδιαίτερη περίπτωση. Είναι διαφορετική από τη Μεσόγειο. Είναι άλλη ιστορία. Σε ό,τι αφορά τα έξι παράκτια κράτη, δεν μιλάμε μόνο για τουρισμό, για τις, ε, για τις αλληλευτικές δυνατότητες. Εδώ ο κόσμος ζει από αυτή την ιστορία, ζει από, το, από την αλληλεία. Ε, θα πρέπει να εξασφαλίσουμε λοιπόν το μέλλον του και να βγάζει πραγματικά αξιοπρεπόστα προς το ζήν. Θα πρέπει λοιπόν να λάβουμε υπόψη μας και το περιβάλλον και τις άλλες ιδιαιτερότητες της Μαύρης Θάλασσας. Θα πρέπει να διαφυλάξουμε τα θαλάσσια αποθέματα. Κάποια είδη της Μαύρης Θάλασσας τα τελευταία χρόνια έχουν εξαφανιστεί. Και μάλιστα διάφοροι συνάδελφοι ε, εξέφρασαν την έκπληξή τους που υπάρχουν ακόμα ψάρια στη Μαύρη Θάλασσα. Με αυτή την έκθεση που θα συζητήσουμε και θα υιοθετήσουμε σε λίγους μήνες, ελπίζω, να συνεισφέρουμε κι εμείς για να ρυθμίσουμε τα τεκτενόμενα στη Μαύρη Θάλασσα. Ευχαριστώ τους συναδέλφους από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Γενική Διεύθυνση ΜΑΡΕ, με τους, τους οποίους γνωρίζω καλά. Εκτιμώ τις προσπάθειες που κάνει και η Επίτροπος ε, η κυρία Δαμανάκη και εγώ είχα επαφές ε, με Τούρκους ομολόγους μου στην Άγκυρα καθώς και με Ρώσους ομολόγους μου Και αυτοί σκέφτονται τι προοπτικέ τη Μαύρη Θάλασσα. Δεν μιλάω μόνο για τι αλληλευτικέ προοπτικέ, αλλά γενικά τι οικονομικέ προοπτικέ τη ε, λεκάνη αυτή. Πρέπει να χρησιμοποιήσουμε κάθε ευκαιρία για να υπογράψουμε μια συμφωνία με αυτέ τι χώρε. Και νομίζω ότι είμαστε καθοδόν και ελπίζω να υποστηρίξετε τι μελλοντικέ μου προσπάθειες. Σα ευχαριστούμε κυρία Ιώτοβα. Ευχαριστώ και του δύο πυρογνώμους, τον κύριο Κοσποντίνοφ και τον κύριο Ραίκο. Θα ήθελα να καθορίσουμε το χρονοδιάγραμμα που θα ακολουθήσουμε ως εξής. Παρουσίαση του σχεδίου έκθεσης στις 12 Τετάρτου. Συζήτηση των τροπολογιών 31 Πέμπτου. Ψηφοφορία στην Επιτροπή 13 Εβδόμου. Και ψηφοφορία στην Ολομέλεια την πρώτη Ολομέλεια του Σεπτεμβρίου. Περνούμε στο επόμενο θέμα σχέδιο προϋπολογισμού 2012. Η συγγήτρια, η κυρία Ρέιμερς, ακόμη δεν υπάρχει σχέδιο προϋπολογισμού για το 2012 μέσω Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Έχει οριστεί ο γενικός εισηγητής ή γενική εισηγήτρια, σε συγκεκριμένη περίπτωση, την οποία συνάντησε η κυρία Ρέιμερς και θα ήθελε να μας κάνει μία πρώτη παρουσίαση των συζητήσεων που έκανε και των γενικότερων γραμμών της έκθεσης αυτής που αφορά τον προπολογισμό του 2012. Κυρία Ρέιμερς, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ. Εγώ συζήτησα με την κυρία Μπαλζάνη, την εισηγήτρια. Είχαμε μια πρώτη επαφή και μια ανταλλαγή απόψεων. Προς το παρόν πρέπει να σας πω ότι είμαστε στο πρώτο στάδιο της ε, διαβούλευσης. Η έκθεση το κείμενο της Επιτροπής ε, το νωρίτερο που θα το έχουμε είναι 20 Απριλίου. Η κοινή αλλιευτική πολιτική, η μεταρρύθμιση της κοινή ε, αλλιευτικής πολιτικής θα παίξει ένα καθοριστικό ρόλο για το 12. Έχουμε ήδη κάποιες ε, ιδέες για το πώς θα τοποθετηθούμε και βεβαίως σκοπός μας είναι να προωθήσουμε θέσεις όσον αφορά την αηφόρο ανάπτυξη, την προστασία του τομέα της Αλίας. Η κυρία Μπαρζάνη σαφώς και είπε ότι θα κατευθυνθεί προς δύο ε, προσανατολισμούς, στρατηγική 2020 και οι θέσεις απασχόλησης. Εμείς θέλουμε να στηρίξουμε κάποιους στόχους και να θέσουμε προτεραιότητες. Το καλύτερο βεβαίως για μας θα ήταν να διαπιστώσουμε Ποια είναι τα πιλωτικά προγράμματα που πήγαν καλά, τα οποία θέλουμε να διατηρήσουμε και πριν ξεκινήσουμε να προωθούμε νέα πιλωτικά προγράμματα, νέα προγράμματα, υπάρχουν τρία που συνεχίζουν να λειτουργούν και τα οποία θέλουμε να αξιολογηθούν και ε, γι' αυτό ζητώ από όλους τους συναδέλφους ε, που είναι οι δικές σας προτεραιότητες, που είναι τα σημεία τα οποία θέλετε να στήριξουμε και να προωθήσουμε. Πιστεύω ότι όσο πιο ευρεία συμφωνία υπάρχει μεταξύ ημών, τόσο πιο εύκολο θα είναι να προωθήσουμε τα θέματα αυτά. Αυτό που είναι πολύ σημαντικό είναι βεβαίως ο στόλος Όλοι ξέρουμε ότι δεν θέλουμε να, να αυξήσουμε συγγνώμη, το δυναμικό. Το θέμα είναι η ηλικία αυτών των ε, σκαφών. Το θέμα βεβαίως των ε, πολιτικών ε, του εξοπλισμού. Του ζητάμε διαρκώς και περισσότερα όσον αφορά τον εξοπλισμό ασφάλειας, όσον αφορά την αξιοπιστία και την ασφάλεια αυτών των σκαφών, ενδιαφερόμαστε για την ζωή τους, για την υγεία τους, θα πρέπει επίσης να συζητήσουμε και το θέμα των ε, μικρών οικογενειακών ε, εκμεταλλεύσεων, επιχειρήσεων, την ανανέωση του στόλου, παραδείγματος χάριν. υπάρχουν προβλήματα όπως ακριβώς και με τα παλιά οχήματα, ένα παλιό λεωφορείο του οποίου η μηχανή δεν δουλεύει πια, ο κινητήρας πρέπει να αντικατασταθεί, ο νέος κινητήρας καταλαβαίνετε ότι μπορεί να προκαλέσει προβλήματα σε ένα παλιό ε, όχημα. Το ίδιο ακριβώς συμβαίνει και με τα σκάφη αυτά. Θα πρέπει λοιπόν ε, να θέσουμε εδώ κάποιους ε, προτεραιότητες και να προωθήσουμε προτάσεις που να μπορούν να ε, προχωρήσουν και να γίνουν αποδεκτές. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Έχουμε το προσχέδιο προπολογισμού 2012. Δεν έχουμε μπροστά μας δημοσιονομικές ε, προοπτικές, αλλά φέτος φαίνεται ότι θα γίνει και η μεταρρύθμιση της κοινή αλληλευτικής πολιτικής. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε ποιοι είναι οι αντικειμενικοί στόχοι που θέλουμε να ειδοποιήσουμε και τι θέλουμε να κάνουμε κάθε χρόνο. Διότι η μεταρρύθμιση θα ε, απαιτήσει περισσότερα κονδύλια και για κοινωνικούς λόγους και για να υλοποιηθεί και η στρατηγική 2020. Επίσης, το θέμα της έρευνας είναι πάρα πολύ σημαντικό η καταπολέμηση της ε, παράνομης αλίας και ένα, θα πρέπει να γίνει ειδική μνήα, πράγμα το οποίο είναι θέμα δυναμικότητας του ελευτικού μας τόλου, είναι το θέμα της ε, ε, αλίας στην ανοιχτή θάλασσα. Όλα αυτά θα πρέπει να τα εξετάσουμε στα πλαίσια της μεταρρύθμισης. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Έχω μία ερώτηση. Υπάρχει κάποιος εκπρόσωπος της Επιτροπής σήμερα εδώ? Όχι. Θα ήθελα να κάνω ερωτήσεις στην Επιτροπή. Είμαι σκιώδης. Όχι. Να περιμένουμε να εμφανιστεί. Κύριε Σπρέιρα, ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την εισηγήτρια για την ε, παρέμβασή της σε σχέση με τα πιλωτικά σχέδια. Η ομάδα μας παρουσίασε πάρα πολλές φορές τα τελευταία χρόνια σχέδια πιλωτικά για την ε, παράκτια αλληλεία. Από ό,τι κατάλαβα, κανένα από αυτά τα σχέδια δεν εγκρίθηκε. Ίσως θα υποβάλουμε και άλλου τέτοιου είδους προγράμματα. Θα ήθελα να πιστήσω την προσοχή των συναδέλφων σε ένα ιδιάζον θέμα αυτής της μικρής βιοτεχνικής αλίας και παράκτιας αλίας. Νομίζω ότι Βρισκόμαστε σε εξίσου κακή, για να μην πω χειρότερη κατάσταση, με αυτή την οποία αντιμετωπίζουμε το 2008, στην πρώτη κρίση των καυσίμων. Διότι, όπως ξέρετε, τις τελευταίες εβδομάδες υπάρχει αυξητική μεγάλη τάση της τιμής των καυσίμων, του πετρελαίου, και αν δεν υπάρξει κάποια προσαρμογή στις τιμές ή κάποια ε, άλλη προσαρμογή, η τάση είναι να αυξηθεί ακόμη περισσότερο η τιμή τη πετρελαίου. Καταλαβαίνετε πόσο αυτό επηρεάζει την ε, μικρή αλία και την ε, αλία την παράκτεια. Τρομερά προβλήματα. Και νομίζω ότι θα πρέπει να μπορέσουμε να κινητοποιήσουμε μέσα για να βοηθήσουμε αυτόν τον τομέα παρά το γεγονός ότι στο παρελθόν τα πράγματα γίνανε τον καλύτερο δυνατό τρόπο αλλά σε αυτό είναι άλλο θέμα τα μέσα τα οποία χρησιμοποιήθηκαν δεν κατευθύνθηκαν στους κατάλληλους, κατάλληλες για άλλη κατεύθυνση. Αυτό είναι ένα θέμα. Εν πάση περιπτώσει, νομίζω ότι στο εγγύ μέλλον θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε και αυτό θέμα τη ανάγκη ε, ε, εξέβρεση επιγόντων μέτρων για να προσαρμοστούμε σε αυτή την αύξηση. Διότι, όπως σας λέω, φαντάζομαι ότι δυστυχώς φτάνουμε σε μια κατάσταση κρίση πριν να φτάσουμε και στο 2012. Τώρα, σε σχέση με αυτό το οποίο ανέφερε η συγγήτρια. Η υποστήριξη δηλαδή για τον εξυγχρονισμό του ε, αλληλευτικού στόλου. Πιστεύω ότι αυτό είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα και συμμεριζόμαστε το θέμα αυτό. Συμφωνούμε απόλυτα δηλαδή ότι είναι αναγκαίο να μελετήσουμε μέτρα τα οποία θα μπορέσουν να μας οδηγήσουν σε εξυγχρονισμό του αλληλευτικού στόλου, όχι μόνο όπως αναφέρθηκε για λόγους ασφαλείας, αλλά για να γίνει η ελία πιο αποδοτική και από ενεργειακής πλευράς. Μας απασχολεί λοιπόν αυτό το θέμα και νομίζω ότι θα πρέπει να δοθούν κάποιοι πόροι για να βοηθηθεί η βιοτεχνική ελία και παράκτια ελία Επαναλαμβάνω. Ευχαριστώ. Κύριος Κούν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Δεν είμαι ειδικό για θέματα προπολογισμού, αλλά θεωρώ ότι είναι καθοριστικό το θέμα. Πώς δηλαδή στο μέλλον ο προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα οργανωθεί στο σύνολό του, εάν ε, θα συνεχίσει η διαπραγμάτευση μεταξύ κρατών μελών όσον αφορά το 0,3% του ΑΕΠ των κρατών μελών. Αν κοιτάξει κανείς δηλαδή τα 7 επόμενα χρόνια, για τέτοια ποσά μιλάμε. Η Επιτροπή βεβαίως θα απαντούσε καλύτερα την ερώτησή μου. Πόσο θα είναι το ποσό που θα διατεθεί συνολικά στον τομέα της αλίας και κατόπιν ε, ανατομέα κυρία Ράιμστερ ίσως έχει μια γενικότερη εικόνα. Αναφέρεται ένα ποσό σε δισεκατομμύρια. Πώς είναι για τον τομέα μας, πόσα δισεκατομμύρια. Πάντα είναι λιγότερα από αυτά που ελπίζουμε. Και βάσει τι δυνατότητες έχουμε. Ξυγχρονισμός, Βέβαια, δεν πρέπει να συνεχίζουν ε, να χρησιμοποιούνται οι παλιές ε, μηχανές δίζελ. Ε, μιλάμε για πολιτική με περιβαλλοντολογικούς στόχους. Η ουσία όμως είναι κατά πόσο θα μπορέσουμε να χρηματοδοτήσουμε όλα αυτά. Δεν έχουμε αυτή τη στιγμή καμία σιγουριά για χρηματοδότηση. θα ήθελα να πω και εγώ το εξή. Ακόμη δεν έχουμε το προσχέδιο προπολογισμού, αλλά δεν ξέρουμε ποια είναι τα τελικά ποσά. Ούτω ή άλλω πρέπει να πω ότι ποτέ τα κονδύλια για την Ελλήνη δεν ξεπέρνουν το ένα δι. Κυρία Ράιμερ, θέλω να ρωτήσω το εξή. Πώ προβλέπετε να κάνετε την αξιολόγηση των πιλωτικών σχεδίων και των δράσεων προτεραιότητα θα το κάνετε με την ε, Κομισιόν και μετά θα μας ενημερώσετε ή θα έρθει η Κομισιόν στην Επιτροπή και θα το συζητήσουμε το θέμα. Πώς θα ασχοληθείτε διαδικαστικά με αυτό το θέμα. Δεύτερον, εσείς μιλήσατε για την ε, ανανέωση για τον εξυγχρονισμό του ολυφτικού στόλου. Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει διαρθρωτική πολιτική την οποία γνωρίζουμε και η οποία θα αλλάξει με τη μεταρρύθμιση κοινή αλληλευτική πολιτική. Ίσως, δεν το ξέρω, αλλά πρέπει να πω ότι αυτή τη στιγμή έχουμε την πολιτική που έχουμε σύμφωνα με τους κανόνες που ισχύουν και κάθε χώρα έχει τα προγράμματα υποστήριξης ε, και την βοήθεια που παίρνει για τον εξυγχρονισμό για άλλα θέματα. Δεν βλέπω πώ μπορούμε εδώ να αλλάξουμε μέσω του προπολογισμού 2012 αυτή την πρακτική. Διότι ο προπολογισμό του 2012 δεν είναι προπολογισμό μεταρρύθμιση τη κοινή αλληλευτικής πολιτική. Του 2013 θα είναι αυτό τη μεταρρύθμιση. Άρα νομίζω ότι δεν έχουμε τη δυνατότητα αυτή τη στιγμή να κάνουμε τίποτε, δεδομένου ότι οτιδήποτε καινούριο θα πρέπει στα πλαίσια τη μεταρρύθμιση. Άρα δεν βλέπω να προβλέπεται τίποτα το εξαιρετικό για τον προπολογισμό 2012, ε, εκτός από αυτά τα οποία προβλέπονται στα πλαίσια των κονδυλίων που χορηγούνται μέσω του ε, Ταμείου Υποστήριξης της Αλίας. Ή αλλάζουμε τη ε, διαθετική πολιτική μας και το ξανασυζητούμε το θέμα αυτό ευθύς από την αρχή ή δεν βλέπω πώ μπορούμε να κάνουμε κάτι τέτοιο όπω το αναφέρετε Αυτή είναι τουλάχιστον η δική μου άποψη και τα σχόλιά μου μετά την πρώτη παρουσία στην οποία κάνετε. Έχετε το λόγο για να ολοκληρωθεί η συζήτηση του θέματο. Ευχαριστώ. Θα προσπαθήσω να απαντήσω σε αυτά που άκουσα. Κοιτάξτε, ε, είχαμε την ευκαιρία να συζητήσουμε. Μέχρι τώρα δεν υπήρχε συζήτηση. Μας έδιναν ένα ποσό και τίποτα παραπάνω. Για το 12 παραδείγματο χάρη αυτό είναι το ποσό. Άνοιξε λοιπόν μια συζήτηση. Υπάρχει βεβαίω και η δημοσιονομική πειθαρχία η οποία είναι ένα γενικότερο θέμα τη Ευρωπαϊκή Ένωση, όχι μόνο για το δικό μα τομέα. Θα δούμε λοιπόν τι δυνατότητε υπάρχουν. Η γενικότερη κατάσταση από οικονομική απόψεω τη Ευρωπαϊκή Ένωση είναι γνώστη. Η προσωπική μου λοιπόν, αν θέλετε, προσπάθεια, αυτό που θα ήθελα εγώ να δω, να γίνεται είναι τα πιλωτικά προγράμματα, όπως είπατε, να συζητηθούν με την Επιτροπή, με τους σκιώδεις εισηγητές, γιατί είναι σημαντικό να έχουμε μία άποψη ολοκληρωμένη και με συνοχή. Και με αυτόν τον τρόπο να μπορούμε να λάβουμε υπόψη μας όλα αυτά τα στοιχεία στην γενικότερη συζήτηση που έχουμε για τον προπολογισμό. Γιατί εμείς είμαστε ένα μικρό τμήμα του συνολικού προπολογισμού. Θα ήθελα λοιπόν να σας πω σήμερα ότι κατά κάποιο τρόπο έχουμε ξεκινήσει κάποιες σκέψεις, έχουμε κατά νου κάποιες ιδέες για το πώς θέλουμε να προχωρήσουμε, ε, να δούμε τι δυνατότητες έχουμε για το μέλλον, όσο και μικροί να είμαστε να προωθήσουμε κάποιες ιδέες στη συζήτηση για τον προπολογισμό και να δούμε τι μπορούμε να πετύχουμε. Δεύτερον, θα ήθελα επίσης να σας πω ότι στις 20 Απριλίου, όπως σας είπα, θα δημοσιευθεί το έγγραφο της Επιτροπής. 24 Απριλίου πιστεύω ότι θα έχουμε την πρώτη ανταλλαγή απόψεων εδώ στην Επιτροπή Αλίας. Θα δούμε τι αριθμοί μας ε, προτείνονται και τι συγκεκριμένο μπορούμε να προτείνουμε. Εγώ θεωρώ ότι θα πρέπει να θέσουμε τις προτεραιότητές μας. Τι είναι επίγον, τι δεν ανταποκρίνεται σε αυτά που θέλουμε. Έχουμε ένα συγκεκριμένο περιθώριο ελιγμού, αν θέλετε. Αλλά θα πρέπει έτσι κι αλλιώς να περιοριστούμε στις προτεραιότητές μας. Σας ευχαριστώ πολύ. Ολοκληρώσαμε και τη συζήτηση του θέματος αυτού της Δεν θα σας παρουσιάσω το χρονοδιάγραμμα για αυτό το θέμα. Άρα ολοκληρώθηκαν οι εργασίες μας για σήμερα και τώρα θα έχουμε την συνεδρίαση των συντονιστών και κλεισμένων των θυρών. Λύεται η συνεδρίαση για δύο λεπτά. Πρέπει να φύγω από την αίθουσα και αμέσω μετά θα αρχίσει η συνάντηση των συντονιστών.